Je peux vous inviter à regarder... Σας παρακαλώ να καθίσετε. Παρακαλώ. On y va, on y va. Ξεκινάμε. Παρακαλώ καθίστε. Ετοιμαστείτε. Κυρίες και κύριοι, είναι η μεγάλη, η τελευταία μεγάλη ψηφοφορία μας, πέραν της απογευματινής για τα κατεπήγοντα, τελευταία ψηφοφορία για μας, για μένα, Ήθελα απλώς να σας πω και συγγνώμη για τους διερμηνεί που θα πρέπει να το ψηφίσουμε. Χρειάστηκε να ψηφίσουμε 20.690 φορές στο, στην και 35.095 τροπολογίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συνεργασία σας. Να περάσουμε απευθεία στι ψηφοφορίε. Ξεκινάμε με την έκθεση του κυρίου Βούγιανιτ. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση με τσόλα. Και πάλι ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση με τσόλα. Και πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Κράτσα για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Σύνολο του κειμένου. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 CP. Ονομαστική ψηφορία. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 21. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 35. η ψηφοφορία. Ονομαστική. Τώρα έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διάνοντα τη χειρό, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Η συγγήτρια, η κυρία Κράτσα, που βρίσκεται, σα δίνω το λόγο. Ήθελα να... Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για τη συμβολή τους σε αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τη χρηματοδότησή τους ε, και ήθελα να παρακαλέσω να αναβάλουμε την, ε, μην προχωρήσουμε στην τελική ψηφοφορία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Διανάταση τη χειρό λοιπόν. Πρόταση αναβολή. Ε, υπέρ τη αναβολή. Κατά. Αποχέ. Οπότε η ψηφοφορία βάλετε. Περνάμε στην έκθεση τη κυρία Μέσνερ. Πρώτα απ' όλα έχει ζητήσει το λόγο ο κύριο Σλίτερ πριν την ψηφίσουμε. Κύριε Σλίτερ, έχετε το λόγο. Θα Eh, ναι. Υπάρχουν κάποια σφάλματα στη Σουδική εκδοχή του κειμένου. Το είχα πει και τη Δευτέρα κατά την έναρξη τη Συνόδου Λομέλεια. Χρειάστηκα να μιλήσω με του γλωσσομαθεί νομικού και θα πρέπει να λυθούν αυτά τα μεταφραστικά σφάλματα, διότι είναι πολύ σημαντικά και αφορούν την ίδια την αρχή των διαπραγματεύσεων με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό, Πρόεδρε, ήθελα να τονίσω ότι η αγγλική εκδοχή είναι η επίσημη. Σε αυτήν θα πρέπει να βασιστούμε τη στιγμή τη ε, ε ψηφοφορία και μετά θα κάνουν τι απαραίτητε διορθώσει οι νομομαθεί Η νομικοί. Η σουηδική μετάφραση δεν συμφωνεί με την αγγλική πάντω και αυτό να το έχουν όλοι υπόψη του και κατά την ψηφοφορία. Πρόεδρο, ευχαριστούμε για αυτήν την παρατήρηση. Την είχατε ήδη ε, υποβάλει. Οπότε θα φροντίσουμε να υπάρχει και διορθωτικό για τη σουηδική μετάφραση ώστε να μπορέσουν όλοι να κάνουν τη σωστή απαλήθευση εκ των υστέρων. Η συγκεκριά μα, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λόγω ε, αυτών των λάθων ήδη υπήρξε η αναβολή από την Τρίτη για σήμερα και η πρωτότυπη γλώσσα ήταν τα αγγλικά στα οποία διαπραγματευτήκαμε και πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιο είναι το θέμα. Πρόκειται για οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια χωροταξία και μην ξεχνάμε πως έχουμε πάρα πολλές ακτές ε, στην ε, Ευρώπη και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για την παραγωγή ενέργεια ε, κτλ. Αυτό είναι το νόημα αυτή τη οδηγία. Πιστεύω πω οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, γι' αυτό ήθελα να το πω. Μετά τις παρατηρήσεις αυτές ψηφίσουμε για το σύνολο του κειμένου. Υπέρ. 88. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφέ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. 88. Τροπολογία τραν. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Πρόταση νομοθετικού ψήφισματο. Μάλλον πρόταση της Επιτροπής προηγουμένως. Διανάταση της χειρό υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Γκαρίγκα Πολέντο. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και ταπανών. Ξεκινούμε με τροπολογία 20D. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Ένα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε Υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Θα επαληθεύσουμε για την πέμπτη τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Κρίμα. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Διονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Ονομαστική ψηφορία μάλλον. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Αγκρίνεται. 27. Υπέρ. Διονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. Διονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εδάφιο 11. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Θέλετε επαλήθευση. Ωραία. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα της, της παραγράφου ε, της παραγράφου 11. Άρχεται η ψηφορία.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 Άρχεται η ψηφοφορία. Τρίτο τμήμα. Κάνουμε παλήθευση. Πέρα Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 10. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έχετε αμφιβολίες. Να επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε για την 20. η παράγραφο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 19. Ανομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το ψήφισμα υπέρ. Συγγνώμη. Ε, άρχεται. Le Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση ΣΒΑΜ για τις παραβιάσεις των διατάξεων των νομοθεσίας του ανταγωνισμού. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία Εκλού. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίθηκε Έκθεση ΣΤΑΣ Μπλοκ 1, τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπλοκ 2 καταπίπτει. Άρα πρόταση της Επιτροπής στο ΡΕΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τροπολογία 35 ακόμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Έκθεση Προτάσιεβιτς για τις νέες ψυχότροπες ουσίες. Το πακέτο των 48 τροπολογιών της Επιτροπής Λιμπίπερ κατά αποχές εγκρίθηκαν. Τροπολογία 12 της Λιμπε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 47 κατά τμήματα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροποποιημένη πρόταση επιτροπής υπέρ. Ήταν σαφές. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Για το δεύτερο τμήμα επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα του 47. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Πρόταση της Επιτροπής τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Και με ονομαστική ψηφοφορία το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Έκθεση της κυρίας Χιμένεθ Μπεθερίλ Μπάριο. Πρώτα το πακέτο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα επαληθεύσουμε για την 17. Ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε, είχατε δίκιο. Πρόταση της Επιτροπής τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Πέτερλε. Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω. Αλλά να το παληθεύσουμε. 5 λοιπόν, τροπολογία 5, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 5, ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Έξι τώρα. Να σηκώνετε καλά τα χέρια. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλλά δεν είναι σαφές. Ωραία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Να σηκώνετε καλά τα χέρια. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία αριθμό 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίφθηκε ήθελα να πω, ήθελα να πω απορρίφθηκε. Είναι το τελευταίο, ναι. Και ονομαστικά τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης, παρακαλώ. Ψηφίστε. Τι θέλετε, να επαληθεύσουμε. Ωραία, θα επαληθεύσουμε για την τροπολογία 3. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Και τώρα περνάμε στο ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τώρα, προτάσει ψηφίσματο τη Επιτροπή Κρατικών Υποθέσεων για τι θρησκευτικέ ελευθερίε και πολιτισμική πολυμορφία. Έχουμε ένα κείμενο, τη παραγράφου 7, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το ψήφισμα ονομαστικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Υπάρχει διαδικαστικό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για διαδικαστικό. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακόμη μια φορά ψηφίζουμε μια έκθεση μετά και απειλούμε την αντιδημοκρατική Ρωσία. Ε, δεν είναι επί της διαδικασίας λέει η Πρόεδρος. Αλλά μην ξεχνάμε πως η δική σας κυβέρνηση κατοχής Διακόπτη ο Πρόεδρος, δεν είναι διαδικαστικό, συνεχίζουμε τις εργασίες μας και περνάμε σε ανακοίνωση... Α, ότι έχουμε τον κύριο Πίτερ Ποσόμκο, που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεργασίας με την Επιτροπή μας για την Ουκρανία. Χαιρετίζουμε στα θεωρία την παρουσία του. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Περνάμε τώρα. Α, θέλετε το λόγο, κυρία Χάρμς, παρακαλώ. Για διαδικαστικό. Ναι, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι.